πρόσωπο του ΕΛΚ που ήρθα επίση. Δεν χρειάζεται να μπούμε στην ουσία, είναι τεχνικό καθαρά το θέμα, αλλά αν έχετε τυχόν ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Η πρόεδρος, ποιος θέλει να μιλήσει, ο κύριος Φόντεκαμφ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την σαφέστατη θέση του, δεν υπάρχει καμία παρανόηση. Θα ήθελα μόνο να ρωτήσω, ίσως μάλλον την Κομισιόν ερωτώ, ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά το Λίχτενστάιν και την ένταξή του στο Σέγγεν στις χώρες του Σέγγεν. Μας είπε ότι πρέπει να, να γίνει υπογραφή ενός πρωτοκόλου. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Δεύτερη ερώτηση. Λέει εδώ ότι θα υπάρχουν μειωμένα δικαιώματα ψήφου για τους εκπροσώπους της ε, Ελβετίας και της, του Λίχτενστάιν. Θα ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχει ακριβώς αυτός ο περιορισμός των δικαιωμάτων ψήφου. Ε, απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στην Κομισιόν, ρωτάει η Πρόεδρος. Ε, ναι. Ε, ποιος θα απαντήσει από τους δύο εκπροσώπους. Η κυρία Μπαρακόφσκι ένα. Α, α, θα απαντήσει ο κύριος Μπόουενς. Εφόσον βρίσκομαι ακόμα εδώ, Πρόεδρε, θα συνεχίσω εγώ. Ένας φίλος από την Προεδρία που βρίσκεται κοντά μου μου λέει ότι το θέμα αυτό βρίσκεται προς την ολοκλήρωση της εξετασή του από το Συμβούλιο και σύντομα θα υποβληθεί στην κρίση του Κορεπέρ. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε βεβαίω όλα αυτά. Για το δεύτερο ερώτημα, σα ζητώ να συγχωρήσετε, Πρόεδρε. Το συζήτησα με τη συνάδελφο. Δεν άκουσα το ερώτημα το δεύτερο ολόκληρο, αν μπορούμε να το επαναλάβουμε. Κύριε Φαντεκάμπ, θα μπορούσατε να το επαναλάβετε. Πρόεδρε, ναι. Στο σχέδιο γνωμοδότηση από τον εισηγητή μα, λέγεται ότι τα δικαιώματα ψήφου των εκπροσώπων τη ομοσπονδία ε, Ομοσπονδίας της και του πριγκυπάτου του Λίχτενστάιν θα είναι περιορισμένα σε επίπεδο Frontex. Το ερώτημά μου είναι γιατί και τι σημαίνει αυτό. Είναι γιατί δεν έχουν διεθνή ύδατα. Τι νόημα έχει. Ευχαριστώ. Όχι, όχι. Η απάντηση είναι απλή. Η Frontex είναι κοινοτικό οργανισμό. Τα κράτη αυτά είναι, συνεργα... είναι συνδεόμενα κράτη, αλλά δεν είναι κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θεσμικό θα ήταν ανέφικτο να του δώσουμε πλήρε δικαίωμα ψήφου είναι εκπρόσωποι χωρών που αντικειμενικά παραμένουν τρίτες χώρες σε σχέση με τις φορές και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κίνητρο για να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για ένταξη. Κύριε Δεκλέστρετε, να σχολιάσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να υποθεί έχει ήδη καλυφθεί. Ωραία. Έχουμε κλείσει λοιπόν με το σημείο 15 τη ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Συμφωνία επανεισδοχή μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Πακιστάν. Αυτή είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε για το θέμα αυτό. Τον Σεπτέμβριο του 2000 το Συμβουλίο ανέθεσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία επανεισδοχή με το Πακιστάν. Οι διαπραγματεύσει ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2007 και η συμφωνία ξεκίνησε να ισχύει το Σεπτέμβριο του 2008. Και τον Μάρτιο του 2009 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου να περατωθεί η συμφωνία με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου έχει αλλάξει ως προς τη σύναψη, ως προς την ολοκλήρωση μάλλον της συμφωνίας. Πριν θα πρέπει να συγκατατεθεί το Κοινοβούλιο για την ε, περάπτωση τη συμφωνία. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στην, ε, στον εισηγητή, να πω για την προηγούμενη έκθεση του κ. Ντεκλά ότι η υποθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ορίζεται την 3η 11 Μαου το μεσημέρι. Σα θυμίζουμε ότι δεν μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίε για την ίδια τη συμφωνία, αλλά μόνο για το σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματο. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση ΚΛΑΣ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στη συνεδρίαση τη 31η Μαου και 1η Ιουνίου Αυτά ως προς το χρονοδιάγραμμα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σόγκορ. Thank you. I will try to speak in Ευχαριστώ. Θα αποπειραθώ να μιλήσω ουγγρικά. Ε, Εδώ είναι... Υπάρχουν ε, αρκετά ερωτήματα Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα όσον αφορά αυτή την έκθεση. Ελπίζω τα μέλη να έχουν πάρει την έκθεση. όσον αφορά την συμφωνία αυτή επανεισδοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πακιστάν. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν ε, τεθεί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε λάβει ορισμένες απαντήσεις από το Συμβούλιο. Και επί τη βάση αυτών των απαντήσεων μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ακόμα και αν η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει εκδώσει μία σαφή γνωμοδότηση, δεν έχουμε κανένα λόγο να απορρίψουμε εμείς αυτήν την έκθεση. Διότι μετά από εννέα χρόνια δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί γρηγορότερη, ταχύτερη πρόοδο στο Πακιστάν. Και κάτι άλλο. Το Πακιστάν δεν έχει υπογράψει, δεν έχει συνυπογράψει τη σύμβαση της Γενέβης, αλλά έχουν επιτύχει πρόοδο, διότι έχουν γίνει διαβουλεύσεις με τις ε, αρχές του Πακιστάν και πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα νέο Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πακιστάν. Και για να μπορείτε να συγκρίνετε ορισμένα στοιχεία, οι χώρες που έχουν συνυπογράψει τη σύμβαση το 68, όπως η Τουρκία, 1968, όπως η Τουρκία, ε, συμφωνούμε όλοι ότι παρόλο που υπάρχει υπογραφή της Τουρκίας υπάρχουν πολλά θέματα σοβαρά στην Τουρκία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν δεν βλέπω το ότι επειδή δηλαδή το Πακιστάν δεν έχει υπογράψει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα. Ορισμένοι συνάδελφοί μου, φιλελεύθεροι μου έχουν ε, θέσει το θέμα αυτό, μου έχουν ζητήσει να προσέξω πολλά σοβαρά ζητήματα, αλλά δεν ωφελούμε σε τίποτα τους χιλιάδες πρόσφυγους, πρόσφυγες, συγγνώμη, αν αρνηθούμε αυτήν την ε, υπογραφεί αυτή την έκθεση και γι' αυτό υποστηρίζω την υπερψήφιση του σχεδίου εκθέσεως. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Υπάρχει άλλος συνάδελφος, η κυρία Γκυγιόμ και η κυρία Φλόρ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για αυτή τη συμφωνία επανεισδοχής που διαπραγματευόμαστε εδώ και 9 χρόνια, προσθέθηκαν και περίπου άλλες 10 με τις οποίες ασχολήθηκε και το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία αλλά δεν είχαμε καμία ανακοίνωση για αυτές τις ήδη υπάρχουσες περίπου 10 συμφωνίες. Μπορέσαμε επίσης να συζητήσουμε κάποια θέματα με την Επιτροπή πέρσι το, Φεβρουάριο, το, το προηγούμενο Φεβρουάριο δεδομένου ότι είχαμε κληθεί όπως και η ΑΦΕΤ να συζητήσουμε το όλο θέμα, το σχέδιο συμφωνήσεως κατά την άποψή μου περιλαμβάνει και κάποια ερωτηματικά τα οποία δεν ε, μπόρεσαν να εξελιχθούν και ακόμη και μετά τη συνάντηση με την Επιτροπή. Όταν πρόκειται για προσφυγή στο Λεσέπασε το ευρωπαϊκό, ε, τι γίνεται δεδομένου ότι το Πακιστάν είναι μια ιδιαίτερη χώρα. Αυτή τη στιγμή της ε, συζήτηση πρέπει να σας πω ότι πάρα πολύ, έχω πάρα πολλούς ενδιασμούς αναφορά αυτά τα θέματα. Και πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Για κάποιους λόγους που ανέφερε, και αυτό δεν με εκπλήσει ο εισηγητής, το θέμα της στήρησης κάποιων διεθνών συμβάσεων δεν βλέπω να υπάρχουν και βεβαίως αναφέρομαι στη Σύμβαση της Γενέβης, την οποία αναφέρατε και εσείς. Δεν νομίζω ότι έτσι με μία μόνο κοντιλιά μπορεί κανείς να αποκλείσει αυτή την σύμβαση της Γενέβης και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα την αξιολόγηση τέτοιου είδους συμφωνιών. Γι' αυτό μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι πρέπει μέχρι τον φθινόπωρο να έχουμε αξιολόγηση για να αρθούν κάποιες απορίες και να έχουμε μία καλύτερη εικόνα του πώς συμπεριφέρονται οι χώρες αυτές στα πλαίσια των συμφωνιών επανεισδοχής. Το λέγω αυτό πριν να υπάρξει οριστική συμφωνία και υπογραφή γιατί θα θέλαμε να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε κυρία Φλότ. Ε, εκ μέρους της κυρίας η οποία είναι εισηγήτρια στην Επιτροπή ΑΘΕΤ για το σχέδιο αυτό έκθεσης, να πω ότι θα στήσει στους συναδέλφους της Επιτροπής της να απορρίψουν την πρόταση για διαφορετικούς λόγους που ήδη έχουν παρουσιαστεί στην Επιτροπή μας. Η συνεδρίαση άλλωστε που οργάνωσε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με τους επικεφαλείς διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κατόρθωσε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας είναι η ολοκλήρωση συμφωνίας επανεισδοχής με το Πακιστάν και μεταξύ των μετρών που προτείνονται θα ε, ληφθούν και μέτρα κατά το Αφγανιστάν. Μιλάμε για επιστροφή Αφγανών και εδώ βεβαίως προκύπτουν αρκετές σοβαρές απορίες για το εύρος του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας αυτής. διότι ως μη Πακιστανοί ω τρίτη μπορεί να θεωρηθούν και πολίτε που έχουν φτάσει απευθεία στο, ε, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαιως αυτό αφορά και την Τουρκία. Εδώ επηρεάζεται και η Συμφωνία Επανεσδοχής με την Τουρκία η οποία δεν δέχεται να διαπραγματευτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπραγματεύσει παράλληλε και με άλλε χώρε πηγέ τη μετανάστευση και των ανθρώπων αυτών, ε, όπω το Πακιστάν. Εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρξουν καταστροφικέ συνέπειε από την χρήση των αδειών κυκλοφορίας. Και σε περίπτωση που δεν παρουσιάζονται έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα από το... δεν παρέχονται μάλλον έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα από το κράτος του Πακιστάν. Αυτό είναι μια διαδικασία που απίστευτο να πιστέψει κανείς ότι υπάρχει. Εδώ πηγαίνουμε σε διαδικασίες της δεκαετίας του 90 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους απάτριδες Αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα σε καταχρήσεις ε, ανυπολόγιστες δεδομένη και τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν βεβαίω. Είναι και άλλα τα τεχνικά ερωτήματα που γύρει η συμφωνία αυτή. Και πραγματικά από τεχνική άποψη η ποιότητα τη συμφωνία μου φαίνεται ιδιαίτερα αμφίβολη. Από πολιτική άποψη πολύ ανέντιμη ε, έναντι μια χώρα όπω η Τουρκία που κοιτάζοντα με τέτοια συμφωνία έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι εκείνη μπορεί να βρεθεί στη θέση να δεχθεί στο έδαφος της ε, Πακιστανούς και Αφγανούς που βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι πέραν των γενικών επεκτητικών σχολείων που πολλές φορές είναι και τεκμηριωμένα κατά της ε, συμφωνία αυτή, ιδίω στον τρόπο αξιολόγηση και ιδίω στην την αρχή τη μη επαναπρόθεση και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν για όλου αυτού του λόγου ηχηρά να απορρίψουμε την πρόταση αυτή και να εξασκήσουμε την αρμοδιότητα που έχουμε αναλάβει ω βουλευτέ σε ένα τέτοιο ζήτημα. Θα πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο πραγματικά να σταθμίσει του τι είδου εντολή θα πρέπει να δώσει μελλοντικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέτοιου είδου έργο. Ευχαριστούμε, κυρία Γκρίσπετ, για να κλείσουμε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο ως και συγκήτρια της ομάδας των φιλελευθέρων και δημοκρατών και λαμβάνοντας αφορμή από την παρέμβαση της κυρίας Φλότρο θα επαναλάβω και εγώ το εξή σημείο Αυτά που προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν προβλέπουν μόνο διαδικασία συναπόφαση, αλλά και αυξημένη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των υποχρεώσεών μα. Έτσι λοιπόν, όπω τελευταία ομιλήτρια, εκ μέρου τη ομάδα μα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με του υπολείπου βεβαίω συναδέλφου για το θέμα αυτό, αλλά να εκφράσω κι εγώ την ανάγκη να φανούμε ιδιαίτερα συνετοί. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν αρκεί. Όπως είπε και ένας συναδελφός μας, ήταν ε, πολύ χρονοβόρα η διαδικασία διαπραγμάτευση τη συμφωνία αυτή. Όμω, στα δικά μου τα μάτια αυτό δεν αποτελεί καθόλου εγγύηση ποιότητα. Το αντίθετο θα έλεγα. Το γεγονό ότι το κράτο αυτό σήμερα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση τη Γενέβη, αυτό το γεγονό θα πρέπει να μα κάνει ακόμη περισσότερο επιφυλακτικού. Η ασφάλεια, η τήρηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προφύλαξη των ε, προσωπικών δεδομένων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε τέτοιου είδου καταστάσει. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε συνεχώ κατά νου. Το Πακιστάν είναι ένα κράτο όπου η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το λιγότερο επισφαλής. Είναι μάλλον ε, ηρωνικό να το λέμε έτσι. Ιδίω η κατάσταση των γυναικών και των παιδιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και νομίζω ότι πολλοί ήμασταν αυτοί που λάβαμε πληροφορίε από διαφορετικέ πηγέ, ιδίω από μη κυβερνητικέ οργανώσει, όπου απεικονιζόταν ή τουλάχιστον επισημάνονταν, επισημένονταν η κατάσταση των Πακιστανών που επαναπροωθούνταν προς τη χώρα τους, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, διότι νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για λόγου σύνεση είναι να φανούμε ιδιαίτερα επιφυλακτική τη στιγμή τη ψηφοφορία. Τα μέλη τουλάχιστον τη ομάδα μου δεν θα αντιταχθούν στην ε, σύναψη συμφωνίας. Δεν είναι επί της ουσίας η αντίρρησή μας. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο στη σχέση μας με το χώρα αυτή για τις συνθήκες επανεισδοχής, όμως επίγει και θα πρέπει και λόγω των νέων μας ευθυνών να αποσπάσουμε μια πραγματική αξιολόγηση της χρήσης των δεδομένων. Και να ξεφύγουμε από αυτή τη δικαστική ομίχλη στην οποία έχουμε περιέλθει. Τη νομική μάλλον ομίχλη στην οποία έχουμε περιέλθει. Ως προς τους όρους και την αξιολόγηση των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που αφορά μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ κυρία Γκρίσμπεκ. Θα καλέσω τώρα πρώτα το Συμβούλιο, μετά την Κομισιόν, να απαντήσει στα σε ορισμένε από αυτέ τι επιφυλάξει που εκφράστηκαν από όλα τα μέλη. καταρχά ο κύριος Μπουργκος από πλευρά Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλούμε για το θέμα αυτό της Συμφωνίας Επενδυσοχής. Ελέγχθη αυτό από πολλούς συναδέλφους. Από το 2000 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι σε κοινοτικό επίπεδο να ολοκληρωθεί τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να πω ότι από την οπτική πλευρά του Συμβουλίου για την μεταναστευτική πολιτική οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι κλειδί πολύ σημαντικές. Μέχρι τώρα είχαν γίνει διμερείς συμφωνίες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και το πλεονέκτημα της κοινοτική, αν θέλετε, ε, σύναψης τέτοια συμφωνίας μας επιτρέπει όχι μόνο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί αλλά και να ασκούμε έλεγχο από κοινοτικής πλευράς πολύ καλύτερα και κυρίως να λαμβάνεται υπόψη μετά από τέσσερι ισχύ του συνθήκη Λισαβόνα και η άποψη του Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Εμεί ε, υποστηρίζουμε την αξιολόγηση τη Κομισιόν και ζητήσαμε και στο Κοινοβούλιο την ε, εξουσιοδότησή του για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην σύναψη αυτή τη συμφωνία. Άκουσα ποιες είναι οι ανησυχίες που εκφράστηκαν και έχουν εκφραστεί και γραπτός. Είναι το θέμα της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν και στις γειτονικές του χώρες. Γι' αυτό το θέμα θα ήθελα να πω ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι το τελευταίο βήμα στην μεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή, κάποιος επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του εάν είναι σαφές ότι δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν η αίτηση ασύλου ή διεθνούς προστασίας του απερίφθη, εάν απεδείχθη ότι δεν έχει το δικαίωμα να έχει άδεια παρανομής στις χώρες μας για λόγους προστασίας, αν δεν, έχει, αν δεν δικαιούται άδεια παραμονής, την οποία έχει ζητήσει εκ των προτέρων, και εάν είναι σίγουρο ότι γίνεται ε, σεβαστή η αρχή της μίας παναπρόθεσης. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν αυτές τις αρχές. Και όπως σας είπα, το τελικό βήμα, το τελικό στάδιο είναι η Συμφωνία Επανεισδοχής. Εάν αποσταλεί κάποιος λοιπόν στο Πακιστάν, σημαίνει ότι το κράτο μέλος που έχει κάνει όλα αυτά τα διαβήματα που προανέφερα τα έχει φέρει σε πέρας ώστε αυτό το στάδιο να είναι το τελικό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι με τέτοιου είδους συμφωνίες και με όλες τις άλλες κοινοτικές συμφωνίες είναι να χειριστούμε κατά κάποιο τρόπο τη μοίρα των Πακιστανών υπηκών και των Αλαδαπών. Και κυρίως πιστεύουμε ότι κυρίως αφορώνται από αυτή τη συμφωνία οι Πακιστανοί. Τώρα, όσον αφορά υπηκόους τρίτος χωρών, είναι σημαντικότατη η αρχή της μη επαναπρόθεσης, την οποία θα πρέπει να σεβαστεί οποιοδήποτε χώρα πριν να φτάσει σε αυτό το τελευταίο στάδιο της επανεισδοχής. Γι' αυτό θα θέλαμε η συμφωνία αυτή να μπορέσει να υπογραφεί με το Πακιστάν, δεδομένου που σας λέω είναι το τελικό στάδιο όλων αυτών των διαδικασιών. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπόργος. Ο κύριος Ντεμπράουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα παρέμβω εδώ για να στηρίξω τον κύριο Μπούργος και τα όσα είπε εξ ονόματος της Προεδρίας. Το ζήτημα των συμφωνίων επανεισδοχής είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμελείται. Πρέπει να έχουμε την απαραίτητη σύνεση, όπως αυτή με την οποία θέλει το Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα. Όμως, συμφωνίε επανεισδοχής δεν πρέπει να θεωρούνται συμφωνίες που δεν είναι τέτοιε. Δηλαδή, οι συμφωνίε επανεισδοχής είναι συμφωνίε απλής διοικητική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και τρίτη χώρα. Αυτό εξηγεί βάσει ποιες διαδικασίες και με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί μια επιχείρηση επιστροφής και επαναπατρισμού στην ε, εν λόγω τρίτη χώρα των εθνικών της υπηκών ή κάποιων υπηκών τρίτης χώρας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι η Συμφωνία Επανεισδοχής δεν λέει τίποτα, δεν είναι αυτός ο σκοπός της, για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το κράτος μέλος λόγου χάρη που θα εφαρμόσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής θα λάβει απόφαση επιστροφής και θα ασκήσει μέτρο απομάκρυνσης. Τα στοιχεία αυτά τα καλύπτει οδηγία επιστροφής τα οποία έχουν, έχει υιοθετηθεί με την διαδικασία της συναπόφασης και ελπίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι οι συμφωνίες επανεσδοχής αφήνουν άθικτη και θα δείτε ότι σε όλε τι συμφωνίε επανεισδοχή υπάρχουν παρόμοιε διατάξει. Αν καλά θυμάμαι, νομίζω θα τη βρείτε σε αυτή τη συμφωνία στο άρθρο 15, αν δεν απατάει η μνήμη μου. Στη συμφωνία λοιπόν με το Πακιστάν, αφήνουν απολύτω άθικτη, έλεγα, τι υποχρεω... υποχρεώσει και των κρατομελών και των τρίτων χωρών. Τα μέτρα του διεθνού δικαίου, τα μέτρα του εφαρμοστέου δικαίου, και του κοινοτικού δικαίου στην προκειμένη περίπτωση για τα κάτι μέλη δεν αλλάζουν. Και αυτό ισχύει για κάθε κείμενο συμφωνία επανεισδοχή. Αυτό βεβαίω αφορά ιδιαίτερο στην αρχή τη μη Νόρε φουλμό. Η αρχή αυτή έχει ενσωματωθεί στη συνθήκη, ανέκαθεν αποτελούσε τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου και εφαρμοζόταν σε περιπτώσεις κοινοτικού δικαίου ασύλου ε, και ιδίως για αιτήσει ε, ασύλου που απορρίπτονταν. Όλες οι περιπτώσεις όμως απομάκρυσης καλύπτονται και πάλι από την οδηγία επιστροφών. Εδώ αναφέραμε την ανάγκη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει πλήρης διατάξεων στη συμφωνία με το Πακιστάν που διευθετούν το όλο ζήτημα για την προστασία των ανταλλασσόμενων δεδομένων. Επίσης, ε, έγινε αναφορά για το σημείο των αδειών κυκλοφορίας, ε, το των κοινοτικών των της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Αυτό δεν θίγεται στη συμφωνία με το Πακιστάν. Η χρήση τέτοιων αδειών κυκλοφορίας δεν προβλέπονται. Επίσης καταλαβαίνω την ανησυχία κάποιων βουλευτών της Επιτροπής σας διότι πράγματι η έννοια της κοινοτικής άδειας είναι έτσι και κάτι πολύ εξειδικευμένο και ίσως και λίγο παροχημένο λόγω των σημερινών εξελίξεων. Εν προκειμένου, αυτό που συμβαίνει στις συμφωνίες αυτού του είδους, όταν αναφερόμαστε σε κοινοτικές άδειες αυτό που συμβαίνει είναι ότι το έγγραφο αυτό δεν χορηγείται στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, που καταλαβαίνουμε ότι δεν αποδέχεται έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρχή εκτός της επικρατείας του και είναι ένα ad hoc ταξιδιωτικό έγγραφο, ένα συνοδευτικό έγγραφο που περιορίζεται απλώς στα όρια των συμφωνιών αυτού του είδους. Έτσι γίνονται τα πράγματα και αυτό είναι και αντικείμενο των διαπραγματεύσεών μας. Τώρα για την αίτηση για αξιολόγηση. Σίγουρα και τεκμηριωμένη είναι και κατανοητή. Γιατί όμως χρειάζεται η αξιολόγηση, θα ρωτήσει κανείς. Γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου τα διαστήματα, τις διάρκειες για τις οποίες μιλούμε. Το ανέφερε και ο συγκεκριτής σας. Η εντολή ήταν μια από τις πρώτες εντολές που ανατέθηκε. Από το 2000 μάλιστα. Όμω δεν ξεκινήσαμε ευθύ αμέσω τι διαπραγματεύσει, παρόλο που η εντολή δόθηκε τόσο νωρί. Ούτε βεβαίω ήταν απλέ οι διαπραγματεύσει και εύκολε. Να τονίσω λοιπόν ότι το ουσιαστικό που μας ενδιαφέρει για τις περισσότερες συμφωνίες επανεισδοχής που έχουμε ως τώρα είναι ότι εντός, μάλλον πρόσφατα σχετικά όλες ε, περατώθηκαν και πρόσφατα τέθηκαν και σε ισχύ. Αυτή η διαδικασία που αφορά τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο έχουν να κάνουν με το ότι υπάρχει περιθώριο σημαντικό για πληροφόρηση, για ενημέρωση, για να υπάρχουν πορίσματα αξιόπιστα και για τα σημεία που ανέφεραν σήμερα οι βουλευτές της Επιτροπής σας, ώστε η αξιολόγηση να είναι χρήσιμη, επικοδομητική και πλήρης και να μπορούμε να αντλήσουμε και διδάγματα για το μέλλον. Αυτό, Πρόεδρε, σημαίνει ότι για να είμαστε χρήσιμοι και στο Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορούμε να φέρουμε σε αίσιο πέρα σε αυτήν την αξιολόγηση ακόμη, σήμερα, ούτε να την ε, τεκμηριώσουμε αρκετά. Η Επιτροπή λοιπόν θα συμφωνήσει εδώ με την Προεδρία του Συμβουλίου και θα ευχαριστήσει την συγκεκριτή, την σας, τον συγκεκριτή σας μάλλον για την στήριξή του προς την απόφασή μας που θα επιτρέψει την σύναψη της συμφωνίας, αλλά καταλαβαίνουμε ταυτόχρονα το θέμα είναι ευαίσθητο. Είμαστε λοιπόν πρόθυμοι να επανέλθουμε το φθινόπωρο σε αυτή τη συζήτηση, οργανώντας μια γενικότερη, ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων με συμμετοχή και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα για τι συμφωνίε επανεισδοχή, του αντικτύπου του και των πρακτικών που ακολουθούνται σε αυτέ. Ευχαριστούμε, κύριε Ντεμπράουερ. Έχοντα ακούσει τη συζήτηση, έχω την εντύπωση ότι είναι για θεμελιώδου σημασία η αξιολόγηση τελικά. Θα ζητήσω τώρα από τον συγκεκριτή, τον κύριο Σόγκορ, να ολοκληρώσει και από ό,τι καταλαβαίνω την πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα την έχουμε στην συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στο τέλος Μαΐου, σωστά. Διορθώστε με αν έχω σφάλει. Μάλλον έχω δίκιο. Κύριε Σόγκορ. Ευχαριστώ. Να επαναλάβω την άποψη των συναδέλφων μου και να πω ότι είναι σημαντικό το πώς αντιλαμβανόμαστε τις εξελίξεις της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν και σε άλλες τρίτες χώρες. Η συμφωνία ωστόσο αυτή έχει μια πολύ σημαντική συνιστόσα. Προστατεύει τους Ευρωπαίους πολίτες. Διασφαλίζει ένα καλό επίπεδο ασφάλειας. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί επιστροφή κάποιου προσώπου, ανάλογα με την, την αποστολή που έχουν αναλάβει όμως και μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Πολλές φορές λοιπόν είναι δύσκολη η επιστροφή τέτοιων ατόμων ή ομάδων ατόμων στις χώρες ε, προέλευσής τους, εάν δεν υπάρχουν συμφωνίες επανεισδοχής. Μπορώ να δώσω πολλά παραδείγματα, όπως της Τουρκίας ή της Κίνας η Κίνα, η οποία προσχώρησε στην Σύμβαση της Γενέβης το 1982 και τον Νοέμβριο το 2002 επρόκειτο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους Κινέζους. Υπήρχε διαπραγματευτική εντολή. Όμως τον Ιούλιο το 2009 μόλις τότε ξεκίνησαν οι πρώτες διαπραγματεύσεις. Για την ώρα καμία συμφωνία δεν έχει υπογραφεί. Η προσχώρηση στη Σύμβαση της Γενέβης δεν προσφέρει καμία εγγύηση ότι θα περατωθεί και η εξέταση μιας συμφωνίας επανεισδοχής. Εάν μάλιστα δείτε τον ε, παγκόσμιο χάρτη, εκτός από τη Μογγολία, οι περισσότερες χώρες που δεν έχουν υπογράψει την ε, Σύμβαση της Γενέβης είναι χώρες μουσουλμανικές στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Ή χώρε όπου η χωρες οπου η πλειοψηφια του πληθυσμού είναι μουσουλμανική συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας. Εν κατακλείδη λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι παρατείνοντας την ε, σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με καταστάσεις όπου και το Πακιστάν τελικά θα στραφεί κάπως εναντίον μας και θα ε, αποδυναμώσουμε έτσι και τα υπόλοιπα επιτεύγματά μας ως τώρα έχοντας την άρνηση, την απόρριψη μιας συμφωνίας. Πιστεύω ότι τα Υπουργεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λογικά θα σταματήσει να λειτουργεί στο Πακιστάν, όμως θα πρέπει και εμείς να ολοκληρώσουμε αυτή την τόσο δυσχερή διαδικασία. Η πρόεδρος θα έλεγα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Πακιστάν και τους κατοίκους του και, όχι, και σε δεύτερο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωράμε στο 17 επέκταση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγια 2003 2003-109 στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Όπως και με άλλα ντοσιέ που συζητήσαμε σήμερα, αυτό καταρχάς συζητήθηκε υπό τη διαδικασία διαβούλευσης όμως το Συμβούλιο δεν ε, επέτυχε ε, μία συμφωνία πριν από την 1η Δεκεμβρίου και την θέση ενισχύει της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και θα ζητήσω από την Κομισιό να μας δώσει μία σύντομη ανάλυση, ανασκόπηση μάλλον, του θέματος ε, και της ιστορίας αυτής της οδηγίας. Και εν συνεχεία η, η κυρία Γκάς θα μας ενημερώσει και εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θυμίσω το ιστορικό της πρότασης αυτής. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι οι συνθήκες εντό των οποίων οι πολίτες τρίτων χωρών εφόσον ε, είναι κατεστημένοι επί μακρά διάρκεια ε, επικράτεια μελών καλύπτονται από την οδηγία που εγκρίθηκε το 2003 για το καθεστώς του κατοίκου μακράς διάρκειας. Από τότε οι δικαιούχοι της διεθνούς προστασίας αποκλείονται από το πεδίο αυτής της οδηγίας. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε δικαιούχοι επικουρικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2007 υπέβαλε πρόταση παράταση της οδηγίας αυτής, διότι αναγνώρισε το κενό και ήθελε και να σεβαστεί μια δήλωση που είχε κάνει από κοινό με το Συμβούλιο την εποχή της υιοθέτησης της οδηγίας του 2003. Δήλωση που έλεγε ότι θα συμπληρωθεί το νομικό πλαίσιο ώστε να προστατεύεται οποιοδήποτε κάτοικος μακρασδιακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παράταση, διεύρυνση αυτή της οδηγίες είναι σημαντική για το σύστημα, το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, διότι θα παράσχει νομική βεβαιότητα στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και σε ό,τι αφορά την παραμονή του σε ένα κράτος μέλος και έπειτα θα επιτρέψει και καλύτερη ενσωμάτωση των προσφύγων και των ε, δικαιούχων επικορικής βοήθειας στην κοινωνία των κρατών μελών τροποποιήσεις λοιπόν που προτείνει η Επιτροπή σκοπέχουν ε, σύντομα να εξισώσουν τους κατοίκους μακρασδιαρκές με όλους τους υπόλοιπους νόμιμους κατοίκους της επικράτειας των 100 μελών. Συγκεκριμένα, επιτρέπει να λάβει κανείς το καθεστώς κατοίκου μακράς διαρκείας στο κράτος μέλος που έχει χορηγήσει καταρχάς το καθεστώς προστασίας. Έπειτα, επιτρέπει την ε, μετακίνηση της ε, έδρας κατοικίας σε άλλο κράτος μέλος και την απόκτηση καθεστώτος κατοικού μακριτζερικίας σε αυτό το δεύτερο κράτος μέλος υπό τις, υπό την ίδιες προϋποθέσεις με τους άλλους ε, πολίτες τρίτων χωρών. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη να δώσω κάποια παραδείγματα προϋποθέσεων που απαιτούνται για να λάβει κανεί το καθεστώς κατοίκου μακρά στο κάτω μέλο που χορήγησε αρχικά την προστασία. Πρώτον, ο πρόσφυγας ή ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κάποια κατοικία νόμιμη σε ένα μέλο για τα προηγούμενα πέντε χρόνια, ότι έχει σταθερά και μόνιμα έσοδα, εισόδημα αρκετό για να καλύψει τις ίδιες ανάγκες του και αυτές της οικογένειάς του, να είναι ασφαλισμένο ε, για ασθένεια και εφόσον η εθνική νομοθεσία το απαιτεί, να μην αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και τάξη σε αυτό το κράτος μέλος. Διευκρινίζω ότι η πρόταση αυτή λαμβάνει υπόψη και την αρχή που έχουμε συζητήσει στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την ιδιαίτερη κατάσταση των προσφύγων ή των ατόμων που έχουν λάβει επικουρική προστασία, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η αρχή της μη επαναπρόθεσης, τον όρο φουλμό. Όπως το είπατε, το Συμβούλιο έχει εργαστεί σκληρά ως το τέλος του 2008 για το θέμα αυτό, αλλά δεν πέτυχε να συναυθεί συμφωνία. Είχαμε σχεδόν την ομοφωνία όλων βάσει της συμβαστικής λύσης της Γαλλικής Προεδρίας, όμως στο πλαίσιο μάλλον εξαιτία της νομικής βάσης του άρθρου 63 που αναφέρατε κι εσείς, στην τρίτη του παράγραφο και στην τέταρτη παράγραφό του, νομική βάση περί μετανάστευσης, βάση λοιπόν αυτής της, εξαιτίας αυτής της νομικής βάσης απαιτεί το πλήρης ομοφωνία. Κάτι που δεν πετύχαμε. Από την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμβαστική λύση που είχε εξευρεθεί επί Γαλλικής Προεδρίας, με την σχεδόν τέλεια ομοφωνία τηρούσε τα, και σεβόταν τα σημεία κλειδιά της πρότασης της Επιτροπής. Από την πλευρά του το Ευρωκοινοβούλιο είχε σε γενικές γραμμές στηρίξει την πρόταση της Επιτροπής με την έκθεση του Απριλίου 2008 και έτσι δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τις τωρινές προσπάθειες του Κοινοβουλίου να αναθερμανθούν οι συζητήσεις για το ζήτημα, να βρούμε μια λύση σε συνεργασία με το Συμβούλιο και αυτό γιατί από την θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα και μετά, ελπίζουμε ότι γρήγορα θα μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ω συνήθω, η Επιτροπή παραμένει στη διάθεσή σα. Και ιδίω στη διάθεση του εισηγητή, του κ. Μωράη, για οποιαδήποτε διευκόλυνση. Ευχαριστούμε. Ε, um, Ευχαριστώ, Σοφή και ευχαριστώ και την Κομισιόν για την ε, ανασκόπηση αυτού του ντοσιέ. Δεν θα επαναλάβω ε, αυτά τα οποία έχουμε ήδη πει γιατί είναι και το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. <laughs> Σε ευχαριστώ Σόφη για όλα αυτά που είπες και σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Είναι ένα, ένας από τους πολλούς φακελούς ε, που είχαν συζητηθεί πριν από την θέση ενισχύ της Λισαβόνας, της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, αυτό που πρέπει να επιτύχουμε βεβαίως είναι αυτό που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, μια σωστή, μια καλή πολιτική ασύλου. Και γι' αυτό πρέπει να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα παροχής ασύλου. Ο Μάρτιν Μπρούερ προσπάθησε να περάσει την πρόταση αλλά δεν επέτυχε ομοφωνία στο Συμβούλιο και δεν επετέχθη συμφωνία τότε. Τώρα έχουμε μια εντελώ διαφορετική κατάσταση όπου δεν απαιτείται ομοφωνία αλλά επίσης υπάρχει βεβαίως το ενδεχόμενο αυτό να πέσει στη Βελγική Προεδρία και έτσι να διευκολυνθεί η κατάσταση και να υπάρχει θετική αντιμετώπιση στο Συμβούλιο. Εγώ συμφωνώ ε, το με το ότι θα πρέπει να επεκταθεί η νομική ε, βεβαιότητα, η νομική ασφάλεια και να ε, εξεταστούν οι περιπτώσεις ατόμων μετά από πέντε χρόνια νόμιμης ε, διαμονής. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή έναν απολύτως ικανοποιητικό μηχανισμό ανάληψης ευθυνών ε, και ένα βέλτιστο σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση αλλά επιδιώκουμε συνέχεια τη βελτίωση. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε κριτήρια διαμονής, εθνικά κριτήρια ε, και να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο συμβιβαστικό κείμενο του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν ακόμα κρυμμοί ζητήματα. Έχουμε κάνει τις πρώτες μας επαφές με τη Βελγική Μελλοντική Προεδρία. Το σχέδιο εκθέσεως θα είναι έτοιμο Ιούνιο-Ιούλιο και αν συμφωνούν και οι σκιώδεις εισηγητές θα συναντηθούμε τον Ιούνιο για να συζητήσουμε το θέμα, αλλά είμαι γενικά αισιόδοξο ότι θα περάσει αυτή η πρόταση. Very good. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο. Δεν βλέπω το όνομά σας. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε το όνομά σας. Έχετε το λόγο πάντως. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση της ε, επιμέσης πρώτας και θα ήθελα το σύνολο των επιφυλάξεων του Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου να τις αναφέρω και θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Είναι πρωταρχή σημασία στα κράτη-μέλη όταν θα πρέπει να πάρουν την απόφαση εάν θα χορηγήσουν την, ε, την κάρτα διαμονής στον καθένα να δουν κάθε κατάσταση χορηγή χωριστά και να δουν αν ε, ε, πληρούνται κάποια άλλα κριτήρια της ιατρικής ε, κάλυψης, της εργασίας κτλ. Τώρα, το θέμα της απόφασης της απομάκρυνσης από το δεύτερο κράτος μέρος είναι κάτι το χωριστό. Θα πρέπει όμως το πρώτο κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την ε, προστασία την διεθνή να μπορεί να χορηγεί κάποιες αποδείξεις στις ε, νέες διατάξεις θα πρέπει να δούμε τι γίνεται για την ε, οικογενειακή επανένωση. Υπάρχει αυτός με το οποίο το Συμβούλιο. Δεύτερον, τα πέντε χρόνια νόμιμης διαμονή σε μια χώρα, τι γίνονται. Είχαμε ζητήσει από την πρώτη αίτηση μέχρι την πραγματική αίτηση τα χρόνια αυτά να μετρηθούν στα πέντε χρόνια νόμιμης αίτησης. Προτείνει η Κομισιό το ίμιση των ημερών ε, να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό. Δεν Πρόκειται για αυτό το οποίο είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ερώτημά μου είναι ποια είναι η θέση του Συμβουλίου λοιπόν όσον αφορά τον υπολογισμό των πέντε ετών νόμιμης παραμονής. Τι συμβαίνει τουλάχιστον το μισό και ποιος είναι ο νομικός ορισμός που δίνεται σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, είσαστε πάρα πολύ σύντομοι και ακριβείς. Το Συμβούλιο ακόμη για αυτό το θέμα δεν έχει λάβει το λόγο. Κύριε Μπούργο θέλετε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ε, ελέγχθη πολλές φορές εδώ, το Συμβούλιο δεν κατέληξε συμφωνία για την, με το κείμενο της Επιτροπής. Αλλά χρειαζόταν ομοφωνία για να πάρουν απόψη παρά το ότι είχαμε μια κάποια πλειοψηφία. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα με την ενισχυμένη πλειοψηφία θα είναι πολύ πιο εύκολο ίσως να καταλήξουμε συμφωνία. Στα τελευταία κείμενα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο, όντως, ο υπολογισμός του χρόνου για την αναγνώριση αυτού του καθεστώτος ήταν ο μισός χρόνος από τη στιγμή της ε, αίτησης προστασίας μέχρι τη χορήγησή της. Όλα αυτά βεβαίως για να μετρηθούν τα πέντε χρόνια. Αυτό συμφωνήθηκε πλειοψηφικά στα τελευταία κείμενα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχαν ε, διαφορές ή διαφοροποιήσεις. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτηση της κυρίας Βουλευτού σωστά, ούτως ή Σας ευχαριστώ κύριε Μπούργκος. Πριν να επανέλθω στον εισηγητή, μήπως θέλει η Κομισιό να προσθέσει κάτι. Η κυρία Γκά, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι. Κλοντ, θέλεις να συνοψίσεις. Είμαι ευτυχής. Θα ξαναρχίσουμε τη συζητήση τον Ιούνιο, όπως σας είπα. Εάν μπορούμε να τηρήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες και τα πέντε χρόνια, είμαι πολύ ευτυχής. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα. Εκτός αν κάποιος έχει να προσθέσει τίποτα άλλο υπό τα διάφορα, τότε κλείνει, λύεται η συνεδρία.